δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την προετοιμασία της ε, κορυφής της ζώνης ευρώ. Μου λένε ότι πριν ξεκινήσει η συζήτηση υπάρχει μια ε, διαδικαστική πρόταση του κυρίου Γλέζου. Έχετε το λόγο κύριε Γλέζου. Θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ότι πέρα από όλα τα άλλα που γίνονται εδώ υπάρχει ένα αγωνιώδες ερώτημα και στο Κοινοβούλιο και σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους πολίτες της. Τι Ευρώπη θέλουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη των λαών ή μια Ευρώπη των μονοπωλίων και του κεφαλαίου Θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών και της λαϊκής κυριαρχίας ή θέλουμε μια γερμανική Ευρώπη ή μια ατλαντική Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη ισότιμη με ισότιμα μέλη. Θέλουμε μια Ευρώπη αυτόνομη, ανεξάρτητη, αυτοδιοικούμενη και όχι υποτελεί στις Ηνωμένε Πολιτείες ούτε με το εμπορικό ούτε με το στρατιωτικό ΝΑΤΟ θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι στην πατρίδα μου την Ελλάδα υπάρχει, υπάρχουν στρατιωτικές sí. βάσεις Κύριε Γκλέζο, παρακαλώ, αυτό δεν είναι διαδικαστικό το θέμα. Ε, είναι δικαίωμά σας να μιλήσετε μεν, αλλά εγώ θα πρέπει να δώσω συνέχεια στην ε, ε, συνεδριασή μας και θα σας δώσουμε σε έφθετο χρόνο το λόγο. Τώρα μιλάμε αποκλειστικά για την προετοιμασία της συνάντησης κορυφής της Ευρωζώνης. Εξ ονόματος Συμβουλίου, ο Ιταλός Υπουργός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω μέρος στη συζήτηση αυτή που συνεκλήθη η συνάντησή μας η προβλεπόμενη ήδη από τον μήνα Αύγουστο ξέρετε θα ήθελα να πω ότι μια συζήτηση επί της ουσίας για τη συνάντηση κορυφής της ζώνης ευρώ είναι κάτι το πρόωρο σέβομαι πάντα φυσικά τις απόψεις σας αλλά να διευκρινίσω ότι δεν ήταν κάτι το επίσημο και δεν έχει ακόμα ε, καθοριστεί η ημερήσια διάταξη. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση επί της ουσίας του θέματος αυτού τον μήνα Οκτώβριο όμως όταν θα έχουν προχωρήσει τα προπαρασκευαστικά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η προετοιμασία της ζώνης ευρώ είναι κάτι το οποίο ανήκει στον πρόεδρο της, δηλαδή τον κύριο Βαν Ρόμπαϊ, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, και όχι τόσο της Ιταλικής Προεδρίας. Υπό το φως αυτών των σκέψεων λοιπόν και χωρίς να θέλω να προκαταλάβω ε, κάποια ημερήσια διάταξη θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Γενικά θεωρώ ότι η ζώνη ευρώ μπορεί να αξιολογήσει με θετικό τρόπο την ε, έλλειψη ε, όθησης προς την ανάπτυξη που επαληθεύθηκε πρόσφατα σε ένα πλαίσιο, σε ένα κλίμα χαμηλού πληθωρισμού. Εμείς πρέπει να επανέλθουμε στην πορεία αυτή και η στρατηγική μας θα πρέπει να βοηθήσει την εκκίνηση εκ νέου της ζώνης ευρώ, μια πολιτική σταθμισμένη ανάμεσα στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτή πρέπει να είναι η βασική μας προτεραιότητα και όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτό περιμένουν και αυτό αξίζουν. Αυτό σημαίνει ότι ο σωστός συνδυασμός πολιτικών που εφαρμόζονται στις χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ θα αποδώσει. Θα πρέπει εμείς να συντονίσουμε τις διαφορετικές μας πολιτικές αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά μας στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να φέρουμε τα δημοσιονομικά μας σε αηφόρα, σε εισαγωγικά επίπεδα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του χρηματοπιστωτικού τομέα, να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία μέσω των επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι τα πεδία στα οποία θα πρέπει να δράσει η κοινότητα και τα κράτη-μέλη. Η Ιταλική Προεδρία προσπαθεί να διασφαλίσει τον συντονισμό και σε νομοθετικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν πολλές πρωτοβουλίες από το Eurogroup, τον Πρόεδρο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πακέτο μέτρων ανταποκρινόμενοι στο ευρύτερο δημοσιονομικό πλαίσιο, μακροοικονομικό πλαίσιο. Έχει μεγάλη σημασία περιοδικά να ελέγχουμε εμείς τα βήματα προόδου τα οποία συντελούνται. Είναι θεμελιώδες αν θέλουμε εμείς οι στρατηγικές οι οποίες έχουν καθοριστεί να είναι σωστά στοχοθετημένες και στραμμένες προς το μέλλον. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ε, αντίστοιχοι των αναγκών και των ε, προσδοκιών και να καταπολεμήσουμε την κατάρα της ανεργίας. Νομίζω ότι η στρατηγική που ακολούθησε μέχρι τώρα η ζώνη ευρώ είναι μια σωστή. Νομίζω όμως επίσης ότι μπορεί να υπάρξει μια κάποια βελτίωση της πολιτικής αυτής. Νομίζω ότι και στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό μπορούμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Είμαι έτοιμος λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας και να λάβω υπόψη μου επίσης και τη τεχνογνωσία και τις αρμοδιότητες τις οποίες έχετε επιδείξει ότι μπορείτε να ασκήσετε σωστά. Ευχαριστώ κύριε Ντελαβέντοβα. Ο κύριος Κατάινεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να σας παρουσιάσω την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της ε, Ευρωζώνης της 24 ε, Οκτωβρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακόμα βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο, οπότε αναμένω τις απόψεις σας σήμερα για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ευημερία για τους πολίτες μας. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μεγάλες ε, προκλήσεις που υπογραμμίζουν το ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε εύρωστη ανάπτυξη και δουλειές στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Ε, στο άτυπο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ την προηγούμενη εβδομάδα στο Μιλάνο συζητήσαμε πολλά ζητήματα με τους Υπουργούς Οικονομικών. Στο μέλλον όμως θα απαιτηθεί μια κοινή δέσμευση της Κομισιόν των κρατών μελών Η πρώτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων εταίρων. Η πρώτη προτεραιότητα το φθινόπωρο αυτό είναι να στηρίξουμε τις επενδύσεις. Η Ευρώπη έχει πολλά να προσφέρει όσον αφορά την καινοτομία, την το εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και την επιχειρηματικότητα. Για να μεταφραστούν όλα αυτά σε νέες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να προωθήσουμε τι επενδύσει και από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εργαζόμαστε σε ένα συνολικό σχέδιο που θα αντιμετωπίζει και τις δύο πτυχές της υπόθεσης. Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι κοινή. Στο εθνικό επίπεδο, χώρες με μεγάλα πλεονάσματα ε, ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο κυρίως στην έρευνα, την ανάπτυξη και τις υποδομές στο πλαίσιο των δημοσίων δαπανών. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι ευρωπαϊκοί πόροι όπως ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Χρειαζόμαστε επίσης έναν εύρωστο τραπεζικό τομέα και χρηματαγορές για να υπάρχει χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία. Το δεύτερο είναι βεβαίω οι μεταρρυθμίσει που θα απελευθερώσουν το δυναμικό που υπάρχει. Αλλιώ δεν θα έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και δουλειέ. Το θέμα δεν είναι να διαλέξουμε μεταξύ μέτρων της πλευράς της ζήτησης ή της προσφοράς, χρειάζονται και τα δύο. Επίσης, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί το βιώσιμο του κράτους πρόνοιας. Καμία χώρα δεν εξαιρείται από την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Κάποιες βεβαίως βρίσκονται σε πιο πιεστική θέση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο που υπάρχει αποτελεσματικότερα για να υιοθετηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι κανόνες μας ε, δεν εμποδίζουν τις χώρες να μεταρρυθμιστούν. Κάθε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα χωρών που έχουν υιοθετήσει σημαντικές μεταρρυθμίσει. με παράλληλα με μεγάλες ε, δημοσιονομικές προσαρμογές. Υπάρχει όμως ακόμα δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο διακυβέρνηση που έχουμε αποτελεσματικότερα. Τρίτον, πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο των βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών για χάρη και των μελλοντικών γενεών. Τα επιτόκια οπωσδήποτε δεν θα παραμείνουν τόσο χαμηλά για πάντα και μόλις αρχίσουν να ανεβαίνουν το δημόσιο χρέος θα γίνει πιο ακριβό και θα απαιτεί μεγαλύτερο κομμάτι των δημοσίων δαπανών και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Οι πιο ευπαθείς χώρες εδώ πέρα θα πληγούν δυστυχώς περισσότερο από τυχόν νέα στάθεια στις χρηματαγορές. Γι' αυτό απαιτούνται σοβαρές επιλογές. Βλέπουμε πως η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών έχει επιβραδυνθεί και τώρα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των δημοσίων δαπανών. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά πρέπει να γίνουν οικονομίες, αλλά υπάρχει πάντα δυνατότητα επιλογής. Η μείωση των δαπανών αντί για την αύξηση των φόρων και η μείωση των δαπανών που είναι περισσότερο λειτουργικέ και δεν αφορούν το μέλλον είναι νομίζω ο λογικότερο τρόπο. Επίση, μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση μπορεί να ωφελήσει αυτού που χρειάζονται κοινωνική στήριξη και να βοηθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασία μέσω τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματο. Όπω δήλωσε το Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα χρειάζονται περισσότερε προσπάθειε για να μειωθεί το φορολογικό βάρο επί τη εργασία. Ταυτόχρονα πρέπει να αναρωτηθούμε το τι είναι αυτό που δεν επιτρέπει τις Ιδιωτικέ επενδύσει στην Ευρώπη. Το επιχειρηματικό κλίμα στην εσωτερική μας αγορά πρέπει να είναι ευνοϊκό για εταιρείε που επενδύουν. και καινοτομούν και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επανέρχομαι έτσι στις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για ανάπτυξη στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή όμως παρεμποδίζεται από διάφορα δρεωμένα, συμφέροντα και γραφειοκρατικά εμπόδια. Κάποιες χώρες έχουν υπερβολικά πολύπλοκα φορολογικά σύστηματα και άρα μεγάλη γκρίζα οικονομία. Αυτό σημαίνει αναπόφευκτα αλλαγές που δεν σημαίνουν μόνο νέο τρόπο σκέψης αλλά και κάποια δυσάρεστα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Μαγική λύση δεν υπάρχει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα βρούμε ε, κάποια λύση στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και σε τελική ανάλυση όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Θα περάσουμε τώρα στον κατάλογο των ομιλητών. Θα ξεκινήσουμε με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Μπάλτς. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τάχθηκε σαφώς υπέρ του Συμφωνίου Ανάπτυξης και Σταθερότητας και εμείς το χαιρετίζουμε. Κάποια κράτη-μέλη τώρα ζητάνε κάποια ευελιξία. Αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων. Δηλαδή ευελιξία υπάρχει ε, και δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς. Αλλά υπάρχει πάντα συνδεδεμένη με κάποιες προϋποθέσεις με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ε, την υλοποίηση αυτών, όχι μόνο την υπόσχεση μεταρρυθμίσεων. Αυτό ισχύει για μεγάλες και για μικρές χώρες, γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν πλέον να κλείνουν τα μάτια μπροστά στην ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Οι συστάσεις αναχώρα της Κομισιόν και του Συμβουλίου των Υπουργών περιέχουν μια αναλυτική παρουσίαση του τι πρέπει να γίνει και πρέπει να εφαρμοστούν. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις είναι η βάση του να βρουν ένα έφορο έδαφος οι επενδύσεις. Και η σωστή εφαρμογή του εξαπλού και του διπλού πακέτου νομίζω θα δείξουν μια πολιτική η οποία είναι υπεύθυνη απέναντι στους πολίτες μας και στις μελλοντικέ γενναίες. Κάτι το οποίο νομίζω έχει αποδείξει πολλές φορές η οικονομική ιστορία, καθώς δεν είναι δυνατόν να πούμε πως η ανάπτυξη θα βασίζεται στον δανεισμό. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είμαστε υπέρ του συνεχούς δανεισμού. Πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας μας, να ενισχυθούν έτσι οι επιχείρησεις μας και οι πολίτες μας οι οποίοι θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον από οικονομική σκοπιά. Και θα πρέπει ακριβώς να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε σταθερότητα και κυρίως περισσότερη ανάπτυξη και αηφορία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάλτς. Θέλετε να απαντήσετε σε μια μπλε κάρτα κύριε Μπάλτς. Ναι. Ωραία λόγια. Ωραία αυτά που μας είπατε. Ευελιξία για τις ε, χώρες που χρωστάνε, να μην δανειστούμε άλλο. Σε ποιο πλανήτη ζείτε εσείς. Βλέπετε πως τα μέτρα που λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται αποτυγχάνουν παταγωδός στις χώρες της κρίσης. τάπε και ο κύριος Επίτροπος. Ε, δηλαδή αυτή την επιτυχία των μέτρων που μας είπατε, πού την είδατε, πόσο καιρό θα παίζουμε πια αυτό το παιχνίδι. Εάν με είχατε ακούσει σωστά κυρία Φωνστόρχ, θα με είχατε καταλάβει κιόλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είπα σαφώς, ε, χαλαρώστε να συζητήσουμε θέμα. Είπα σαφώς πως υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας εντός των υφιστάμενων κανόνων. Δεν έχω πρόβλημα λοιπόν με το να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες αλλά μην τους παραβιάσουμε. Και δεν ζούμε σε κανέναν άλλον πλανήτη. Αγωνιζόμαστε καθημερινά και θα χαιρόμουν και τα άλλα κόμματα εδώ πέρα να κάναν το ίδιο, να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, να φέρουμε επενδύσεις στην Ευρώπη. Και όταν λέτε πως δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ναι, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως σε κάποιους τομείς ε, όπου ήταν τα πράγματα δύσκολα, έχουμε κάποιες πρώτες ε, αχτίδες ελπίδας τουλάχιστον. Παρακαλώ να προσέχετε το χρόνο σας, γιατί όσο περισσότερο χρόνο χρησιμοποιείτε, τόσο λιγότερο θα μιλήσουν οι επόμενοι. Γι' αυτό παρακαλώ θα με αναγκάσετε να είμαι κι εγώ πιο αυστηρός όταν υπερβάλλετε. Ελπίζω να το κατανοήσετε αυτό. Εξ ονόματος τώρα της Προοδευτικής Συμμαχίας και της Σοσιαλιστικής Ομάδας, ο κ. Ροντρίγης. Η κυρία, συγγνώμη, Ροντρίγης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κατάινεν, πιστεύω πραγματικά και η ομάδα μου επίσης ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνει ήπειρος με μέλλον, με ευημερία με ορίζοντα ευημερία όπου θα υπάρχουν νέες δεξιότητες, νέα ανταγωνιστικότητα και νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει αυτό στην Ήπειρό μας. Παρόλα αυτά, η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή ανάπτυξη και αποτελμάτωση. Ακόμα και ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού υπάρχει και χάνουμε πολλές καλές θέσεις εργασίας. Η ανεργία μας είναι πολύ ψηλή και ο ρυθμός ανέχειας επίσης. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Εμείς εκλεγήκαμε για να διασφαλίσουμε πραγματική αλλαγή στην Ευρώπη. Εκλεγήκαμε για να διασφαλίσουμε ότι η κύρια προτεραιότητά μας θα είναι η ανάπτυξη, η επένδυση και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε όμως πραγματικές λύσεις και μέχρι τώρα οι λύσεις που προτείνονται από την Κομισιόν δεν δουλεύουν. Αυτό είναι φανερό. Εσείς τονίζετε κυρίως τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Εμείς πιστεύουμε ότι όντως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις όχι όμως μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στην παιδεία και στο σύστημα καινοτομίας και πολλές άλλες. Εκτός από αυτά όμως πρέπει να έχουμε μια νομισματική πολιτική που να υποστηρίζει την ανάπτυξη και μια συντονισμένη οικονομική πολιτική με βάση τη ζήτηση και πολλές περισσότερες επενδύσεις που να προσβλέπουν στο μέλλον. Αυτό σημαίνει βέβαια και ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση που θα συνοδευτεί από την Τραπεζική Ένωση να συνοδεύεται και από την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία. Έχετε μπλε κάρτα, θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πραγματικά συγκλονίστηκα με αυτά τα οποία είπατε, πώς διαβάσατε διάφορες γενικολογίες, διάφορες κοινοτοπίες που δεν έχουν κανένα νόημα. Τα θέλετε όλα ταυτόχρονα και δεν σας ενοχλούν οι αντιφάσεις που υπάρχουν στο λόγο σας. Θέλετε μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων και ταυτόχρονα δημοσιονομική εξυγίανση. Θέλετε να μειώσετε τα χρέη και να μειώσετε και τους φόρους. Και πολιτική ζήτηση και μέτρα προώθησης της ε, προσφοράς. Ε, δεν γίνονται όλα μαζί. Αυτά που είπατε τα θεωρώ νομίζω ένδειξη της απελπισίας ε, με την οποία εμφανίζεστε εσείς υποψήφιος για το σημαντικότερο οικονομικό χαρτοφυλάκιο. Μιλήσατε για το ότι ο δημόσιος πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η Ευρωζώνη μπήκε σε κρίση ακριβώς επειδή έπεσαν τα επιτόκια στην Νότια Ευρώπη ε, όταν υιοθετήθηκε το ευρώ και ξεκίνησε εκεί πέρα ο δημόσιος τομέα να κάνει πολύ περισσότερες επενδύσεις που δεν ήταν αποδοτικές και που δεν ε, είχαν κανένα έσοδο και καμία απόδοση. Σήμερα είναι τέσσερις φορές χαμηλότερα τα επιτόκια. Άμα δεν επενδύουν οι ιδιώτες το κάνουν γιατί δεν θα αποδώσουν τίποτα αυτές οι επενδύσεις. Και αν δεν επενδύουν γι' αυτό τον λόγο οι ιδιώτες πρέπει να βρούμε την αιτία. Είπατε πως πρέπει τα ζητήματα αυτά να τα δούμε στο υψηλότερο επίπεδο. Το υψηλότερο επίπεδο πρέπει να το δούμε στους ειδικού. Ειδικοί οικονομολόγοι, νομπελίστες έχουν πει πως δεν θα βγει η Ευρωζώνη από την κρίση με μια τέτοια Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούκε. Κοιτάξτε έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Κύριος Δεσεντιούτς έχει ζητήσει και αυτός να κάνει μια ερώτηση προς την κυρία Ροντρίγες. αλλά ξεκίνησε πρώτος ο κύριος Λούκε. Γι' αυτό θα ακούσουμε. Τώρα δέχεστε κυρία Ροντρίγες τη δεύτερη ερώτηση. Ήθελα να σας συγχαρώ για τα καλά σας λόγια τα οποία συμμερίζομαι εν πολλής. Ήταν πολύ ωραίο παρέμβαση. Αλλά συμφωνείτε ή όχι ότι ο καλύτερος τρόπος να πραγματοποιηθούν όλα αυτά είναι να αυξηθεί, να προωθηθεί το πνεύμα επιχειρηματικότητας και να ελευθερωθούν οι επιχειρηματίες από το τεράστιο φορολογικό βάρος, με την περισσότερη ελευθερία δηλαδή. Κυρία Ροντρίγκε. Κοιτάξτε, και εμείς φυσικά είμαστε υπέρ του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Αλλά μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις παρόλα αυτά η διευθέτηση των αγορών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Εδώ έχουμε μια διαφορά δηλαδή για μας. Για να επανέλθει η ανάπτυξη και η απασχόληση δεν είναι απαραίτητο να καταργηθεί το ευρώ. Αντίθετα πρέπει να συμπληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση για να δοθεί ευκαιρία σε όλες τις χώρες μέλη να επιστρέψουν στην ανάπτυξη και να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα εργαλεία που διαθέτουμε ήδη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο συντονισμό στην Ευρωζώνη και περισσότερη κοινωνική διάσταση και τέλος να έχουμε μία λογική δημοσιονομική πειθαρχία για να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι αν και έχουμε ίδιο στόχο οι τρόποι για την εφαρμογή τους του είναι διαφορετική. Ευχαριστούμε κύριε Ροντρίγκε, ο κύριος Γίζεκ, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να θέσω ερώτημα με μπλε κάρτα, αλλά να τονίσω μερικά βασικά στοιχεία για τη συζήτηση. Ο ΣΑ, όπω ξέρετε, Δευτέρα προέβλεψε ότι θα υπάρξει ακόμα λιγότερη ανάπτυξη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως και αυτό σημαίνει ότι τα πολύ δύσκολα μέτρα λιτότητα που εφαρμόστηκαν στην Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία είχαν ως αποτέλεσμα στη ζωή των πολιτών ε, αυτά τα αρνητικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι μερικές μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης ετοιμάζονται όπως η Γαλλία και η Ιταλία να εφαρμόσουν, να ζητήσουν περισσότερη ευληγησία στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης θα ακολουθηθούν αυστηρά μόνο από μικρές οικονομίες και θα ερμηνεύονται πιο ευέλικτα από τις μεγαλύτερες χώρες και τις μεγαλύτερες οικονομίες ή μήπως η Κομισιόν έχει σκοπό να εφαρμόσει αυστηρά τους κανόνες της για όλες τις χώρες. Επίσης για μένα είναι ζωτικό για την αξιοπιστία της Ευρωζώνης στα μάτια των χωρών που δεν είναι μέσα στη ζώνη να γνωρίζουν ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλες τις χώρες. Επίσης είναι σαφές ότι οι αποφάσεις της Ευρωζώνης έχουν επιπτώσεις και στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ερωτώ λοιπόν πώς θα διασφαλίσετε ότι η Ευρωζώνη δεν θα παραμείνει ένα απομονωμένο μπλοκ και πώς θα διασφαλίσετε ότι οι χώρες της θα αναλάβουν και τις ευθύνες για τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ για την συνομοσπονδιακή ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχει το λόγο η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι το σύνθημά μας όπως είχε πει και ο Τομάζο Ντελαμπεντούζα απαιτούνται διαφθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές και καταλήγουμε πάντα στην καταστροφή την οικονομική. Η Ευρωζώνη πηγαίνει προς τη διάλυση, δεν υπάρχουν επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας μειώνονται συνεχώς. Απαιτείται μια γνήσια εναλλακτική λύση. Δυστυχώς όμως οι προτάσεις τις οποίες κάνετε δεν αλλάζουν καθόλου. Η λιτότητα δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, η λιτότητα και η δημοσιονομική εξυγίανση από μόνες τους δεν δημιουργούν ανάπτυξη. Έχετε προσπαθήσει επανειλημμένα προς αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες δεν σας πιστεύουν. Είπαμε τα αποτελέσματα της πολιτικής σας είναι καταστροφικά. Η καταστροφή μάλιστα αν μπορώ να το πω έτσι χειροτερεύει από, ε, από τη μία περίοδο στην άλλη. Υπάρχουν διάφοροι φανατικοί υπεφιλελεύθεροι οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν καθόλου κανόνες. Πρέπει να καταργηθούν όλοι οι κανόνες και τότε τα πράγματα θα φτιάξουν. Αυτό είναι πραγματικά ανόητο και εξαντλεί την υπομονή των Ευρωπαίων. Ο κύριος Λάμπερτ, εξ ονόματος των Πρασίνων, Ελεύθερη Συμμαχία. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που με εντυπωσιάζει στις δηλώσεις του Συμβουλίου είναι αυτή η αίσθηση που έχουν τις, ε, το κατεπήγοντος χαρακτήρα. Έχουμε τόσα εκατομμύρια και δεν ξέρουμε ακόμη αν θα γίνει η σύσκεψη κορυφής, πότε κτλ. Είναι όμως κατεπήγον να υπάρξει μια απάντηση. Εγώ αυτά που είπατε τα ακούω εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Δομικές μεταρρυθμίσεις, δομικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή μείωση των δημοσίων δαπανών και μείωση του κόστους εργασίας. Ξέρετε βέβαια ότι αυτές οι δομικές μεταρρυθμίσεις έχουν ως κύριο αποτέλεσμα να πλήττουν τους πιο αδύναμους και όχι τους πιο πλούσιους. Και εμείς είμαστε υπέρ βασικών μεταρρυθμίσεων, αλλά όχι τις, τον, τις ίδιες με τις δικές σας. Θέλουμε να υπάρξουν επενδύσεις, αλλά κατ' εμάς πρέπει οι επενδύσεις να κάνουν την Ευρώπη την πιο οικονομική χώρα στη χρησιμοποίηση πόρων και ενέργειας και αυτό θα αλλάξει πλήρως την οικονομία μας. Πώς θα κινητοποιηθούν ποσά για τις επενδύσεις. Υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν τους χρησιμοποιείτε. Πρώτον, θα συζητήσετε στην Κομισιόν και στο, Σύμβουλο, και στο Συμβούλιο δεσμευτικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη χρησιμοποίηση πόρων. Αν βάλετε λοιπόν δεσμευτικούς στόχους θα γίνει κάτι. Και αυτό δεν το λέω εγώ αλλά οι ίδιες οι επιχειρήσεις αν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες δεν υπάρχουν επενδύσει. Δεύτερον, η κυριότερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι η φορολογική. Σήμερα τα φορολογικά συστήματα είναι και κοινωνικά άδικα και οικονομικά αντιπαραγωγικά και καταστρέφουν το περιβάλλον. Χρειάζεται μια πλήρης αναθεώρηση των φορολογικών συστημάτων. Ξέρω ότι υπάρχει ο κανόνας της ομοφωνίας αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Και τρίτον, όσο θα παραμένει η οικονομία του καζίνου για τις επιχειρήσεις δεν πρόκειται τα ποσά που διατίθενται στην οικονομία να φτάσουν σε παραγωγικές επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το έχει καταλάβει σχεδόν. Πού βρίσκεται η ρευστότητα αυτή τη στιγμή, πού πάει χρηματοδοτεί φούσκες για ακίνητα και κινητές επενδύσεις αλλά όχι δεν επενδύει στην οικονομία είναι εύκολο να κάνει κανείς μεγάλα κέρδη χωρίς να εργάζεται μέσω της σπέκουλας αλλά ε, θέλετε ή όχι επιτέλους να επενδύσετε στην πραγματική οικονομία χωρίς να φέρει το βάρος και ο φορολογούμενος μόνο. Χρειάζονται λοιπόν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά όχι αυτές που προτείνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λάμπερτς. Μια μπλε κάρτα. Δέχεστε την ερώτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Λάμπερτς εγώ είμαι ακαδημαϊκός στον κλάδο της οικονομίας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς οι επενδύσεις στην ενέργεια θα διασφαλίσουν την ευημερία της ζώνης ευρώ. Ένα, δύο, τρία. Να μου πει πώς θα το κάνει. Αγαπητέ ε, κυρία δεν είμαι φοιτητή σας, μπορεί να είστε πανεπιστημιακός, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι επιχειρηματίας ε, εκτός από το ότι έχω διατελέσει ευρωβουλευτής ήμουν επιχειρηματίας. Ε, δεν σας διαφεύγει το ότι όπως είπε ο κύριος Κατάινεν οι επενδύσεις ε, μπορεί να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη ενώ η κατανάλωση από μόνη της δεν θα το καταφέρει αυτό. Στον τομέα της καινοτομίας, ιδιαίτερα στην ενέργεια, δημιουργείται μία κατάσταση δημιουργίας προστιθέμενης αξίας ταυτόχρονα και με ανταγωνιστικό τρόπο πρωτοπορείται σε σχέση με άλλες ζώνες του πλανήτη. Όταν σε κάποια φάση λοιπόν θα πρέπει να μειώσουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε, θα πρέπει εμείς να έχουμε τις λύσεις και να μην αγοράζουμε τις τεχνολογίες που θα απαιτηθούν από τη Βραζιλία και την Κίνα. Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι αποκλειστικά η καταχρηστική ενίσχυση της κατανάλωσης θα μας οδηγήσει στο μαρασμό. Σαφχάουζερ, μπλε κάρτα για τον κύριο Λάμπερτς. Κύριε Λάμπερτς, εγώ φυσικά και δέχομαι αυτά που είπατε για την πράσινη οικονομία και την αηφορία. Αλλά αυτό το οποίο διαρωτώ και θα ήθελα να σας το θέσω σαν ερώτημα είναι να μου πείτε αν δεν αλλάξει η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ή δεν αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα, οι πιστώσεις οι διαθέσιμες να μην πηγαίνουν αποκλειστικά σε τράπεζες αλλά να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα υποδομών όπως ακριβώς το είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αν δεν υπάρξει όμως αυτή η ποσοτική διευκόλυνση των 400 εκατομμυρίων στην αηφόρο ανάπτυξη δεν θα πετύχουμε τίποτα. Κοιτάξτε. Λογικό το ερώτημά σας. Ήδη πρέπει στην Ευρώπη, όχι ίσως στην Αγγλία, στην υπηρετική Ευρώπη να υπάρξει διαφορετική κατανομή των διαθεσίμων πόρων αλλά βλέπω επίσης ότι στην πραγματικότητα η Ευρώπη δεν υποφέρει από έλλειψη ρευστότητας ή κεφαλαίου. Το θέμα είναι πού διατίθενται τα κεφάλαια. Δεν διατίθενται στις επενδύσεις αλλά στην κερδοσκοπία, ιδίω στα ακίνητα. Φαίνεται αυτό στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και αλλού και στις μετοχές. Επομένως το θέμα για μας είναι πού θα αλλάξει, πώς θα, πώς θα μετατοπιστούν, θα μετατοπιστεί η χρήση της υπάρχουσας ρευστότητας και σε ποιο βαθμό βέβαια. Αλλά ήδη να δούμε πού διατίθενται τα μέσα που διαθέτουμε πριν ζητήσουμε πρόσθετα. Η Ευρώπη είναι πλούσια η μην το ξεχνάμε, αλλά τα κεφάλαιά της δεν χρησιμοποιούνται όπως θα έπρεπε. Τώρα θα συνεχίσουμε ο, ο κύριος Βάλι από την ομάδα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος Κατάινεν, ότι χρειάζεται δηλαδή να εξηγιάνουμε το πιστοτικό μας σύστημα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κάποιες σκέψεις. Από ό,τι φαίνεται, εμείς δίδουμε πολύ μεγάλη ρευστότητα στις τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή τους, αλλά αυτά δεν φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Λυπάμαι που δεν είναι ο Ντράγκη εδώ για να μας πει ακριβώς πώς μπορούμε να στοχεύσουμε σωστά τις δυνατότητες ε, ρευστότητας. Εφόσον δεν έχουμε λοιπόν κάποιους συγκεκριμένους στόχους, δεν έχουμε και συγκεκριμένες δεσμευτικές θα έλεγα ε, πρακτικές τις οποίες να ακολουθήσουμε για να ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία. Θα στηρίξω εδώ αυτό που είπε ο κύριος Λάμπερτς. Απαιτείται μια σωστή ρύθμιση των διευκολύνσεων που δίδουμε προς τα πιστοτικά ιδρύματα. Πρέπει να δεσμευτούν ότι οι πιστώσεις που τους δίνουμε θα βγουν στην πραγματική οικονομία, αλλιώς δεν θα βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Για τους ε, μη εγγεγραμμένους ο κύριος Μονό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε ε, σε σχέση με αυτή τη συνάντηση κορυφής. Έχουν γίνει τόσες πολλές μέχρι τώρα. Χωρίς αποτέλεσμα. Από το Μάιο του 10 έχετε προσπαθήσει να σώσετε το ιδιωτικό πιστοτικό σύστημα και τον χρυσόν βού, τον οποίο λατρεύεται, δηλαδή το νομισματικό ευρωπαϊκό σύστημα. Έχετε πάρει μέτρα σύμπτυξης των αμοιβών, των μισθών, των συντάξεων, κάνατε hold up εις βάρος των Κυπρίων κάτι το οποίο δείχνει ότι η νομισματική ευρωπαϊκή ζώνη δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση καλά. Εμείς ε, είμαστε η ζώνη του μηδέν. Μηδέν ανάπτυξη, μηδέν απασχόληση, μηδέν ανταγωνιστικότητα εκτός από τη Γερμανία, μηδέν αύξηση της αγοριστικής δύναμης και τεράστια αύξηση των ελλημάτων. Λοιπόν, παρά τα δώρα που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα πιστοτικά ιδιωτικά ιδρύματα, τα αποτέλεσμα δεν τα είδαμε. Η υπερφιλελεύθερη Ευρώπη δυστυχώς άρχισε να τα χάνει. Και το παράδοξο είναι ότι ο κύριος Γιούνκερ έβαλε ε, για τον έλεγχο των ελλημάτων τον πλέον αποτυχημένο των Ευρωπαίων Υπουργών ως προς το συγκεκριμένο τομέα, τον κύριο Μοσκοβισή. Πού θα πάμε έτσι. Κάθε χώρα στον κόσμο έχει το νόμισμά της στην κεντρική της τράπεζα και τα ελέγχει με τον τρόπο που θεωρεί καλύτερο. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς έχουμε ένα ελληματικό προϋπολογισμό, έχουμε ένα ελληματικό ε, συσχετισμό ε, χρέους ε, γενικά ήδη από το 2003 έχουμε φτάσει σε χρέη απίστευτα υψηλά έχει αποτύχει το ευρώ, έχει αρχίσει και αποσυντίθεται το οικονομικό σας σύστημα και στην ουσία εσείς ζητάτε ε, από ε, τα Υπουργεία Οικονομικών να συμπεριλάβουν και εγκληματικές δραστηριότητες για να αυξήσετε τους αριθμούς όπως την πορνεία, το οργανωμένο έγκλημα κτλ. Ευχαριστώ κύριε Μονό, όχι άλλο. Μία μπλε κάρτα επίσης, πρέσεν. Έχετε το λόγο. Κύριε Μονό, μόλις τώρα μιλήσατε για υπερφιλελεύθερη Ευρώπη. Αναρωτιέμαι σε ποια Ευρώπη ζείτε. Εγώ βλέπω μια υπερσοσιαλιστική Ευρώπη εδώ πέρα κοινωνικοποιούνται τα πάντα. Οτιδήποτε υπάρχει και ακούμε ότι θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο αυτή η κατάσταση. Τι είναι φιλελεύθερο σε όλα αυτά. Αν ήταν φιλελεύθερη εγώ θα την υπερασπιζόμουν. Euh, Κύριε μου, η Ευρώπη δεν είναι απλώς φιλελεύθερη, είναι υπερφιλελεύθερη. Έτσι μας επιβάλλει το διεθνές οικονομικό πρότυπο που εφεύραν οι Αγγλοσάξονες. Φυσικά είμαστε υπέρ του φιλελευθερισμού σε εθνικό επίπεδο και του προστατευτισμού κοινοενουσιακός. Βλέπετε όμως ότι η Ευρώπη χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή από μείωση της αγοραστικής δύναμης και ανεργία. Αυτό, αυτό είναι που σας ικανοποιεί. Δεύτερη μπλε κάρτα. Κύριε Ντελαπίνη. Της κυρίας Ορίστε. Κύριος. Όχι η κυρία. Ακούσαμε πάρα πολύ προσοχή να μιλάτε για την Ευρώπη την οποία δεν επιθυμείτε, για την Ευρώπη που δεν αγαπάτε. Φυσικά και υπάρχουν ευθύνε για την κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα και τις μοιραζόμαστε όλα τα θεσμικά όργανα. Ακούσαμε την κριτική. Προτάσεις όμως, πού είναι οι προτάσεις. Δεν τις ακούσαμε. Κοιτάξτε, γιατί... Κοιτάξτε κύρια μου. Θέλουμε πράγματι την Ευρώπη των εθνών, μια Ευρώπη που να δημιουργεί πλούτο για τους λαούς της και όχι για τις πολυεθνικές και τα ιδιωτικά τραπεζικά συστήματα. Θέλουμε μια Ευρώπη που να κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο και είναι πολύ απλό. Η λύση είναι απλή. Το ίδιο που έκαναν η Αγγλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, η Κίνα. Δηλαδή χρησιμοποιούν το εθνικό τους νόμισμα ως εργαλείο πολιτικής και τα σύνορά τους και έχουν πραγματικά άξιες του ονόματος κεντρικές τράπεζες. Το ίδιο προτείνουμε και εμείς. Το πέρασμα δηλαδή την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα με το ευρώ να παραμείνει απλώς κοινό και όχι ενιαίο νόμισμα. Μόνο έτσι νομίζουμε ότι θα επιστρέψει η ευημερία των λαών. Ε, Τρίτη μπλε κάρτα. Αλλά καθυστερούμε, ε, καθυστερούμε. Όχι, ο επόμενος ομιλητής, κύριος Άγιες από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω την απεσιόδοξη άποψη του προηγούμενου μιλητή σε σχέση με το ευρώ. Εγώ θεωρώ πως το ευρώ θα πετύχει και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή να κάνουμε δύο πράγματα για την οικονομία της Ευρωζώνης και τα 28 κράτη-μέλη. Πρέπει να επιμείνουμε στους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά την σταθεροποίηση του συστήματος της Ευρωζώνης και πρέπει να συνεχιστεί η μείωση των ελλημάτων όπου και αν βρίσκονται. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα που έχει δει τεράστιες μειώσεις στις δαπάνες που είχε και αυξήσεις στους φόρους λόγω της οικονομικής κρίσης. Και όμως στην Ιρλανδία η αύξηση του ΑΕΠ είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη. Οπότε ακόμα και χώρες που κάνουν αυτή την προσαρμογή μπορούν να έχουν ένα παραγωγικό και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης στο μέλλον. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, θεωρώ πως έχει τεράστια σημασία να μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τρελή πολιτική. Έχουμε 11% ανεργία και φορολογούν τον κόσμο μέχρι θανάτου. Δεύτερον, πρέπει να ξαναξεκινήσουν τα δάνεια στις επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν, έχει μειωθούν, όταν έχουν μειωθεί οι επενδύσεις κατά 20% στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκη τα τελευταία 5 χρόνια, πρέπει να ξαναξεκινήσουν οι επενδύσεις. Στο τελευταίο τρίμηνο 50% των επιχειρήσεων απορρίφθηκαν για δάνειο από τις τράπεζες και για χρηματοδότηση. Και συμφωνώ επίσης πράγματι σε μια ενιαία χρήματα αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός τραπεζών. κάτι ακόμα θα πω. 60% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Αμερική είναι από νέες επιχειρήσεις που δεν υπήρχαν το 2008. Το μέλλον της Ευρωζώνης και της Ευρώπης βασίζεται σε ισχυρή ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Χέις. Σας είπα ότι όταν μιλάτε περισσότερο μειώνετε τις επόμενες. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπούλμαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κομισιόν μας λέει πως δεν έχει μαγική λύση. Ε, το ξέρουμε. Αλλά μας το έχει πει και πολλές φορές ήδη. Εντάξει κύριε Επίτροπε, το να μην έχετε μαγική λύση δεν εξηγεί όμως το γιατί ε, εδώ και πέντε χρόνια πηγαίνετε προς τη λάθος κατεύθυνση. Και πρέπει να μας πείτε επιτέλους ε, τι κάνετε όσον αφορά την γενική αντίληψη της οικονομίας σε μια εσωτερική αγορά. Είναι καλύτερη αντίδραση όταν κινούνται τα κράτη-μέλη προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Και δεν μας έχετε πει πώς ακριβώς θα κάνουμε κάτι άλλο πέρα από τις κοινέ περικοπές. Πρέπει να γίνουν επιτέλους και κοινέ επενδύσεις. Επιτέλους, αντελήφθηκε η Κομισιόν πως υπάρχει πρόβλημα και κενό επενδύσεων στην Ευρώπη. Πώς θα γίνει λοιπόν να προχωρήσουμε συνολικά για να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στις επενδύσεις. Αυτά είναι τα σημαντικά. Κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Η Ευρώπη, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι δεν καταλαβαίνουν το τι κάνουμε. Ούτε καν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ε, Φραγκφούρτη. Πρέπει επιτέλους ο κύριος Τράγκη να κάνει κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων. Εντάξει, καλές οι συνοδικορυφείς, αλλά έχει φτάσει στιγμή να κάνουμε και αυτό το οποίο σας είπα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν. Έχετε μία μπλε κάρτα κύριε Μπούλμαν. Δέχεστε την κάρτα. Ναι λέει ο κύριος Μπούλμαν. Ο κύριος Ροπέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Μπούλμαν. Είμαι Λιθουανός και στην Λιθουανία είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να μπούμε στο ευρώ. Ε, ξέρετε ότι για να το κάνουμε αυτό πρέπει να σεβαστούμε και τα κριτήρια του Μάστρεχτ αλλά δεν υπάρχουν κριτήρια που να έχουν σχέση με τον ελάχιστο μισθό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάτι τέτοιο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία υπήρξε. Πείτε μας τι πρόβλημα έχετε. Έχετε ένα πρόβλημα, έχετε ένα πρόβλημα με τη ερμηνεία. Πείτε una tarjeta azul. Ε, trataba de formular la pregunta... Λοιπόν, μπορείτε να θέσετε εκ νέου την ερώτησή σας κύριε Ροπέ, γιατί χάθηκε. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ε, κοιτάξτε, ε, αυτό το οποίο είπα είναι ότι στη χώρα μου, στη Λιθουανία, από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα μπούμε στο ευρώ. Για να το κάνουμε αυτό βέβαια θα πρέπει να σεβαστούμε τα κριτήρια του Μάστερ. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχει η διασφάλιση του ελάχιστου εισοδήματος, του ελάχιστου μισθού, της ελάχιστης αμοιβής έτσι ώστε να φροντίζουμε τους πολίτες μας. Ε, θα ήταν σωστό λοιπόν να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ε, η μπλε κάρτα είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την παρουσίαση την οποία έκανε ο προηγούμενος ομιλητής. Λοιπόν, έπρεπε να κάνετε την ερώτησή σας στον κύριο Μπούλμαν και όχι να την κάνετε στην Επιτροπή. Κύριε Μπούλμαν, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ να απαντήσω στην ερώτηση του συναδέλφου. Κοιτάξτε, ε, πρέπει να σκεφτούμε όμως κάποτε να δούμε και το θέμα του πόσες μπλε κάρτες επιτρέπονται. Να απαντήσω όμως στην ερώτηση. Έχει δίκιο ο συνάλφος. Ε, θα ήταν καλύτερο να ζούμε σε μια Ευρώπη στην οποία θα υπήρχαν σταθερές συμφωνίες ε, για να υπάρχει σε κάθε χώρα ένας ε, ανάλογος βασικός μισθός που θα εξασφαλίζει στον κάθε εργαζόμενο ότι θα μπορεί να ζει από την εργασία του και να μην εξαρτάται από περαιτέρω βοήθεια. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες Παλεύουμε γι' αυτό και συμφωνώ και εγώ και απευθύνω έκκληση σε Κομισιόν και Συμβούλιο να κάνουν μια τέτοια πρόταση να εγκριθεί αύριο διαβοής. Εγώ μη υπέρ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι άκουσα με βάση αυτά που είπατε, δεν έχετε βγάλει και εσείς και η Κομισιόν σημαντικά συμπεράσματα για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση για ποιο λόγο δεν υπάρχει ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή ένωση για ποιο λόγο υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι και θα πρέπει να σκεφτείτε αν το μοντέλο το οποίο χρησιμοποίησε η κομισιόν η ευρωπαϊκή ένωση για την έξοδο από την κρίση ήταν το σωστό και δεν ήταν διότι για το μοντέλο που χρησιμοποιήσατε δηλαδή τη λιτότητα δηλαδή τον αποπληθωρισμό τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά γέμισε η Ευρώπη ανέργους. Δεύτερο, το μοντέλο για την ανταγωνιστικότητα την οποία, το οποίο προωθείται είναι ένα μοντέλο που στηρίζεται στην, στο σύμφωνο για το ευρώ. Δηλαδή στη μείωση των μισθών. Δηλαδή σε ανταγωνιστικότητα η οποία έχει σχέση με το να κινεζοποιηθούν οι μισθοί στην Ευρώπη. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην τεχνολογία, στην οικονομία, και κυρίως στην παιδεία. Αλλά αυτά δεν μπορείτε να τα κάνετε, διότι όταν έχετε μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική, αυτά απαγορεύονται επί της ουσίας. Και δημιουργείται τεράστια προβλήματα, κυρίως στις χώρες του Νότου. Στην Ελλάδα, όπου η πολιτική σας είναι καταστροφική, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, χιλιάδες φτωχοποιημένοι Έλληνες, χιλιάδες κλειστά μαγαζιά, και όλα αυτά από τη δικιά σας πολιτική την πολιτική της τρόικας η οποία έχει καταστρέψει την ελληνική οικονομία. πρέπει να βγάλετε λοιπόν τα απαραίτητα συμπεράσματα και να αλλάξουμε πολιτική διότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση δεν μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα μέλλον σοβαρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και να αναλάβετε και εσείς και η Τρόικα τις ευθύνες για την καταστροφική σας πολιτική στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Μνημονίου. Κύριε Μαριά, έχετε μία μπλε κάρτα. Δέχεστε από την κυρία Γιάκονσάρη. Η κυρία Γιάκονσάρη έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο προς το παρόν η κυρία Γιάκονσάρη. Το μικρόφωνο σας λέει ο πρόεδρος. Μα το έχω ανοίξει, το έχω ανοίξει. Το κόμμα μου είναι το τρίτο κόμμα σε δύναμη στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Επομένως, ή θα έπρεπε να έχετε το θάρρος, κόμμα σας μάλλον, να παρουσιάζετε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Έχετε τις δυνατότητες, αλλά δεν ακούω καμία συγκεκριμένη πρόταση. Ποια είναι η πρόταση της ομάδας σας για να επανέλθουμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση. και από τον κύριο Λούκε και από άλλους. Η βασική αντίληψη είναι ότι με αυτή την πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ευρωπαϊκή ένωση και η πολιτική της λιτότητας δεν μπορούν να δώσουν καμία διέξοδο. δεν μπορούμε να έχουμε μια ευρώπη που έχει γεμίσει ανέργους δεν μπορούμε να έχουμε μια ευρώπη που κερδοσκοπούν οι τράπεζες δεν μπορούμε να έχουμε μια ευρώπη που η ρευστότητα δεν πηγαίνει στην πραγματική οικονομία δεν μπορούμε να έχουμε μια ευρώπη η οποία καταπιέζει τους λαούς του νότου μια ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή έχει διαλύσει όλη την οικονομία στο νότο και έχει γεμίσει ανέργους. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη των εθνών κρατών που πραγματικά μπορεί να δώσει διέξοδο σε αυτή την κατάσταση και όχι μια Ευρώπη των κεντρικών, μια Ευρώπη η οποία καταπιέζει τους ίδιους τους λαούς της. Ο κύριος Γκουερέρο διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, κρίση, η χρήση συγγνώμη, της μπλε κάρτας είναι ένα δικαίωμα του Ευρωβουλευτή και του δίνει τη δυνατότητα να θέσει μια συγκεκριμένη ερώτηση στον προηγούμενο ομιλητή. Εγώ δεν θέτω το θέμα της ανυπαρξίας του δικαιώματος αυτού, αλλά να υπάρξει μια προσοχή παρακαλώ σε σχέση με τη χρήση γιατί ε, κάτι τέτοιο με τον τρόπο που γίνεται δημιουργεί προβλήματα στο χρόνο που έχετε δώσει στις πολιτικές ομάδες, μειώνει ε, τον χρόνο που έχουν ε, οι βουλευτές για να πάρουν το λόγο κανονικά, οι οποίοι έχουν επίσης την ελπίδα να ομιλήσουν και στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye παρακαλώ από το Προεδρείο να είναι πολύ προσεκτικό και επιφυλακτικό και περιοριστικό στη χρήση της λεγόμενης μπλε κάρτας. Κοιτάξτε, ε, προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, η δυνατότητα να τεθούν δύο φορές ερωτήσεις σε κάθε ομιλητή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πράγματι ο χρόνος ε, είναι δικαίωμα το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι βουλευτές. Ο κύριος Παπαδημούλης έχει το λόγο. Ε, κύριοι του Συμβουλίου και της Κομισιόν, ήρθατε μάδια χέρια. Κύριε της Ιταλικής Προεδρίας, πού είναι η στροφή στην ανάπτυξη και οι αλλαγές που μας υποσχέθηκε εδώ τον Ιούνιο ο κύριος Ρέντσι. Κύριε Κατάινεν, πού είναι το πρόγραμμα των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που μας είπε ο κύριος Γιούνκερ. Εδώ εσείς δεν μπορέσατε να μας πείτε ούτε πότε θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής για την Ανάπτυξη. Και την ίδια ώρα η οικονομική ορθοδοξία της κυρίας Μέρκελ αμφισβητείται ακόμη και από τους δικούς της ανθρώπους. Ο κύριος Ντράγκη παίρνει μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, δειλά καθυστερημένα, παρά τα εμπόδια που του βάζει ο κύριος Σόιμπλε Ακόμη και ο ΩΣΑ του νεοφιλελεύθερου κυρίου Γκουρία σας λέει σταματήστε με αυτή την καταστροφική πολιτική, πάρτε μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και στροφή στην ανάπτυξη. Η Γαλλία μονομερός ανακοινώνει ότι μετά από δύο χρόνια θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσει του Συμφώνου Σταθερότητας και εσείς μας λέτε αφόρητες, βαρετές γενικότητες. Την ώρα που υπάρχει υψηλότατη ανεργία, στη χώρα μου την Ελλάδα 30%, 60% στους νέους, την ώρα που η Ευρωζώνη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ύφεση και με τον κίνδυνο του απολυθωρισμού Απαντήσεις περιμένουμε, περιμένουμε από εσά και όχι γενικότητες. Μην μειώνετε και μην κοροϊδεύετε Ναι. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κύριε Κατάινεν, εγώ είχα απογοητευτεί τόσο πολύ από την συζήτηση γιατί το καλοκαίρι μειώθηκε το, ε, συγχωρείτε, επιδεινώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα και βλέπουμε πως δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα. Πάλι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε κάποια μέτρα για να προσπαθήσει να εμποδίσει την κατάρρευση, αλλά εδώ και δύο χρόνια έχουμε την πρόταση των τεσσάρων προέδρων για μια καλύτερη ηγεσία της Ευρωζώνης για περισσότερη ολοκλήρωση, για περισσότερη δημοκρατική νομοποίηση. Δεν άκουσα τίποτα από αυτά. Ανταυτού βλέπουμε μια λογική αναβολής. Είχαμε μια σύνοδο κορυφής αμέσως μετά το καλοκαίρι εκεί πέρα μιλήσανε μόνο για εξωτερική πολιτική και τώρα δεν μπορείτε να μας πείτε καν πότε θα λάβει η χώρα η επόμενη σύνοδος για την ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας και εφαρμόστε επιτέλους τα σχέδια αυτά για να ε, λειτουργήσει και το ευρώ ε, σωστά. Αλλά δεν μας είπατε αυτά, μας είπατε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Οφλίν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Το ευρώ μπορεί να μην έχει καταστραφεί ακόμη αλλά σίγουρα έχει αποτύχει γιατί η βασική δοκιμή είναι εφόσον, ε, το κατά πόσον μια οικονομική πολιτική καταλήγει σε ανάπτυξη και απασχόληση. Η Ιταλική οικονομία, χώρα που ήταν γνωστή για, για τα βιομηχανικά της επιτεύγματα και το design σήμερα δεν έχει καθόλου περισσότερη ανάπτυξη από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Έχει χαθεί μία δεκαετία, δεκαπενταετία. Και ρωτώ κατά είναι γιατί συμβαίνει αυτό στις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης <clears throat> για να προστατευθεί η οικονομία των χωρών αυτών χρειάζεται δικό τους νόμισμα πρέπει να μπορούν να θέσουν και τα επιτόκια τους μόνες τους. Όμως εσείς δεν επιδεικνύεται επαρκή κοινωνική αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζονται αυτοδιαχείριση οικονομική αυτές οι χώρες. Ντροπή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπονάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Κατάινεν. Από αυτά τα οποία μας είπε φαίνεται ότι έχει συνηθίσει να να συνομιλεί με ε, ομολόγους του και στη χώρα του όπως ο κύριος Βικένεν. Εγώ προέρχομαι από τη μικρή πόλη του Μποργοσέζια στο κέντρο της Ιταλίας και κατεβαίνω ε, στην πλατεία την Κυριακή το πρωί και το Σάββατο, βάζω ένα γραφιάκι και ακούω τους συμπολίτε μου. Και τι θέλουν οι συμπολίτε μου, θέλουν λεφτά και κυρίως θέλουν δουλειά. Έχει καταστροφεί η Ευρώπη λοιπόν. Ε, η Ευρώπη δεν δίνει απαντήσεις και ακούω πράγματα τα οποία δεν φαντάζομαι. Εσείς δεν επικοινωνείτε με τον κόσμο αυτό. Μιλάτε μόνο με τους ομολόγους σας, τους γραφειοκράτες και τα μεγάλα παγκόσμια πιστοτικά ιδρύματα. Σκοτίστηκαν για τους πολίτες και τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ντροπή της Ευρώπης και εσείς σε αυτή την πορεία έχετε εντάξει τον εαυτό σας. Ο κύριος Κίρτσος έχει το λόγο, λέει ο πρόεδρος διακόπτοντας τον κύριο Μπονάνο. Ο κύριος Κίρτσος έχει το λόγο. Νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες, διότι χωρίς μεταρρυθμίσεις θα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ιτηθεί οικονομικά από τις Ηνωμένε Πολιτείες, από την Κίνα και από άλλους ισχυρούς ανταγωνιστές. Θεωρώ επίσης ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα ε, είναι αναγκαία διότι διαφορετικά θα πέσουμε σε μια μαύρη τρύπα χρέου, και εμείς στην Ελλάδα πληρώνουμε τώρα όχι τόσο τη δύσκολη πολιτική του μνημονίου όσο τα λάθη που κάναμε τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία 2000-2009 που αντί να προετοιμαστούμε για πρόσθετο ανταγωνισμό στα πλαίσια της ΟΝΕ για παράδειγμα οι Γερμανοί φίλοι μας είχαν το Ατζέντα 2010 εμείς κάναμε παροχές και μας ξέφυγε η δημοσιονομική διαχείριση. Χρειάζεται όμως μια πρόσθετη προσπάθεια, μια δημιουργική σκέψη να συμπληρωθεί ο κορμός της πολιτικής που είναι κατά βάση σωστός. Πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε, πόσο ισχυρό θέλουμε το ευρώ. Θέλουμε πληθωρισμό κοντά στο 0 ή πληθωρισμό κοντά στο 2%. Θέλουμε ρευστότητα, θέλουμε ποσοτική χαλάρωση ή θέλουμε νομισματική ορθοδοξία. Ε, επομένως, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε δεν υπάρχει κανένα αυτοματισμός που να λύνει το πρόβλημα. και τελο θέλω να διαμαρτυρηθώ με διαφορου ευρωσκεπτικιστε ιδιαίτερα του γερμανούς οι οποίοι τελο πάντων κάνουν κριτική στην ελλάδα ζητούν ο Νότο να εγκαταληφθει δεν καταλαβαίνουν ότι άμα πέσουμε εμεί σε ένα μαύρο πηγάδι χρέου, θα παρασύρουμε και τους γερμανούς φορολογούμενους του οποίου υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Η κυρία Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τον Επίτροπο. Η Ευρώπη ακολουθεί την λιτότητα με δογματικό και απόλυτο τρόπο και αυτό έχει οδηγήσει αναπόδραστα στην ύφεση. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όλο και χειροτερεύει ουσιαστικά η κατάσταση. Επί έξι χρόνια ουσιαστικά βιώνουμε μια κρίση. Δεν έχει υπάρξει κάποιο θαύμα. Η κατάσταση δυστυχώς χειροτερεύει συνεχώς. ύφεση και χειροτέρευση επαναλαμβάνω της κρίσης. Ε, η κρίση δεν είναι βέβαια παγκόσμια, δεν είναι σφαιρική. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε που κάποτε ήταν το επίκεντρο της οικονομικής κρίσης έχουν αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό και βγαίνουν από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί, έχει φυσικά βοηθήσει αλλά η ρευστότητα την οποία παρέχει δεν μετατρέπεται σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις Λοιπόν, απαιτείται να αλλάξουμε πολιτική, απαιτείται να διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα έτσι όπως τα κάναμε δεν είναι σωστά. Να μην μείνουμε στα λόγια, να μην μείνουμε παρατηρητές και να προσπαθήσουμε να πάρουμε νέα μέτρα. Η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φοβάμαι ότι δεν θα επιτρέψει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις κατά τη διάρκεια των ακροάσεων έτσι ώστε να μας εμπνεύσει εμπιστοσύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι τα προγράμματα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα γιατί η πραγματικότητα στην παρούσα φάση είναι απειλητική. Τσάνι. Ο κύριος Τσάνι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτοί που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Ρέντσι ε, τους κοροϊδεύουν στην Ευρώπη ο κύριος Κατά είναι να θεωρείται το γεράκι της λιτότητας. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις με το βασίλειο των ζώων. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πρόβατα επισφαγή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα οποία κάνατε μέχρι τώρα όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν καταστροφικά δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση χαρίζοντας 3.000 δις λέει ο μιλητής στα πιστοτικά ιδρύματα. Πότε θα καταλάβετε ότι για να βγούμε από την κρίση δεν χρειάζεται λιτότητα αλλά αλληλεγγύη. Και παρακαλώ μια σύσταση. Η συνάντηση κορυφής ε, για την Ευρωζώνη να την οργανώσετε στις περιφέρειες των μεγάλων πόλεων που δεν έχουν πια ελπίδα, που δεν έχουν πια κατάλληλη κατοικία. Εγώ κάθε εβδομάδα έρχομαι σε επαφή με το λαό. Πηγαίνετε λοιπόν στο σπίτι σας κύριε Κατάινεν, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και αναρωτηθείτε τι κάνω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαριανόπουλος. Ο κύριος Ζαριανόπουλος επαναλαμβάνω. Πρόεδρε, σας θυμίζω ότι κατέθεσα αίτημα στο Προεδρείο σας για να πάρω το λόγο επί σοβαρού διαδικαστικού προβλήματος. Περιμένω μέσα στη διαδικασία να το πάρουμε. Επί του θέματος, Λίγο πριν από τη Σύνοδο της Ευρωζώνης, οι προσδοκίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστω για ανεμική ανάπτυξη, μετατράπηκαν σε φόβο για νέο γύρο βαθύτερης καπιταλιστική κρίση. Οι προβληματισμοί όλων των κομμάτων που υποκλίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την καπιταλιστική ανάπτυξη για κάποια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής με επεκτατική στρατηγική δεν αναιρούν τη δήλωση ενός από τους συζητητές της, του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Ντράκη, που είπε ότι η χαλάρωση δεν θα θίξει τη σιδερένια δημοσιονομική πειθαρχία, τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μείωση των επιτοκίων, η αγορά ομολόγων, οι κρατικές επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο δεν θα αντιμετωπίσουν την ανεργία, δεν θα ωφεληθούν εργαζόμενοι αλλά μόνο τα καπιταλιστικά κέρδη γιατί αυτή η ανάπτυξη στηρίζεται ακριβώς στην ανεργία στη φτώχεια στην κατεδάφιση εργατικών κατακτήσεων της κοινωνικής ασφάλισης των δικαιωμάτων στην υγεία και την παιδεία. τα μέτρα ψίχουλα για την ακραία φτώχεια που εξανεμίζονται από την άγρια αντιλαϊκή φορολογία όχι μόνο δεν δίνουν λύση αλλά ουσιαστικά πιέζουν το γενικό επίπεδο μισθών και συντάξουν σε μια γενική γραμμή φτώχειας με κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων τα προγράμματα απασχόλησης γενικεύουν την προσωρινή ελαστική απασχόληση χωρίς δικαιώματα. κανένα μέτρο δεν μπορεί να σώσει αυτό το σύστημα που σάπισε και δίνει μόνο ανεργία φτώχεια και πολέμους. η μοναδική εγγύηση για τους εργαζόμενους να ικανοποιήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες για μια ανάπτυξη προς όφελός τους είναι η ανατροπή αυτού του συστήματος και της πολιτικής του. Ευχαριστώ, ο κύριος Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και τον Επίτροπο. Είναι προφανές ότι προ στιγμή πρέπει την πρόταση της Κομισιόν να της δώσουμε προτεραιότητα, την ανάπτυξη δηλαδή και την απασχόληση. Βεβαίως, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ιδιαίτερα αυτές της Ευρωζώνης πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα. Είναι μια πρακτική πολιτική πραγματικότητα. Είναι σαφέστατο περισσότερο στην Ευρωζώνη από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά και κάτι άλλο είναι ζωτικό επίσης. Η δημαγωγία είναι κάτι που ακούμε συχνά πια εδώ στην Ολομέλεια. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα πράγματα άσπρο-μαύρο μανιχαϊστικά. Δεν θέλουμε τέτοια λύση. Το Συμβούλιο κάνει προτάσεις με βάση και αυτό τα αποτελέσματα των εκλογών. εκλογών. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις λοιπόν είναι απαραίτητες γιατί χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση. Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες και καιρό είναι πια να τονίσουμε τα δύο αυτά θέματα που οι οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν επαρκώς και με βάση δομικές πολιτικές που έχουμε ήδη συμφωνήσει από κοινού. κύριος Μπαλτιέρη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι βλέπουμε πια με την κρίση ότι αργά αλλά σταθερά βγαίνουμε πια από το τούνελ και ε, αρχίζει να δημιουργείται και κάποια συνένεση ευρεία. Πρέπει να βγούμε πια από τη μονοδιάστατη αντιμετώπιση που είχε πολλές φορές επιβληθεί και να συνδυάσουμε πολλά είδη μέτρων διαχειριστικά, οικονομικά, δημοσιονομικά. Είναι σημαντικό ότι ο Επίτροπος να αναγνώρισε ότι χρειάζονται και επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ότι υπάρχει έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις οι οποίες να είναι στο ύψος των ερωτημάτων. Εμείς θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί ως προς αυτό. Θα επιμείνουμε και για τις επενδύσεις. Απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα 300 δις του κυρίου Γιούγκερ και θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί με αυτά τα οποία είπατε. Και ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, εθνικές επενδύσεις, ευρωπαϊκές επενδύσεις. Βασικά αυτό που θέλουμε είναι fresh money, νέο χρήμα Επίσης τώρα για τις δημοσιονομικές πολιτικές και το θέμα της ευελιξίας. Η ευελιξία δεν είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, η ευελιξία είναι τμήμα του κανόνα. Οι κανόνες ακριβώς ορίζουν την δυνατότητα της ευελιξίας για να αποφευθούν προκυκλικές πολιτικές. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια διορθωτική πολιτική της δημοσιονομικής κατάστασης της Ευρωζώνης, όχι μόνο κάποιων χωρών. Μια λογική συμβατή με την ανάπτυξη που ευνοεί τις διαφθρωτικές αλλαγές γιατί με μεμονωμένες δημοσιονομικές πολιτικές είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Κύριος Βούλφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθώς προετοιμαζόμαστε για τη Σύνοδο Κορυφής ε, της Ευρωζώνης πρέπει να θυμόμαστε κάποια στατιστικά στοιχεία που θα εξετάσουν η πολιτική τη μέρα εκείνη. Το ΑΕΠ έχει αύξηση 0,1% και βεβαίως και βεβαίως το ποσοστό της εργασίας αυτό μειώνεται. Σε χώρες όπως ε, την, εργασία, την Κροατία έχουμε 17% ανεργία 23%, 23-25% στην Ελλάδα. Καλά νέα, έτσι. Όταν ξέρουν πως κάποιοι άλλοι θα κάθονται σε λιμουζίνες, θα πίνουν τη σαμπάνια τους και θα δουν πως θα την περάσουν ακόμα καλύτερα. Αλλά βεβαίως βλέπουμε πως αυξάνεται η ανεργία, μειώνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, αυξάνεται το κόστος της εργασίας. Αυτό το οποίο θα σας έλεγα λοιπόν εγώ κυρίες και κύριοι πως αν κάτι μοιάζει τόσο πολύ με αποτυχία είναι αποτυχία. Αλλά το μόνο που θα μας πούν από αυτή τη σύνοδο είναι «Αχ, επιτέλους ήρθε η επιτυχία». Ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μια παρατήρηση. Πραγματικά προετοιμάστηκε άσχημα αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρουμε καν πότε θα γίνει η σύνοδος ε, κορυφής. Και μιλάμε γενικά. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, να έχουμε έργα τα οποία θα έχουν προταθεί. Και η ε, Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να περιοριστεί στον εαυτό τους. Πρέπει να γίνει ένας κινητήρας της εσωτερικής αγοράς. Ποιοι είναι οι στόχοι μας. Σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, να εφαρμοστούν οι συμφωνίες συντονισμού, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αναμένουμε λοιπόν προτάσεις για το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις και πώς θα οδηγηθούμε σε αυτή την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ποια είναι τα μέτρα. Ναι, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ε, εκπαίδευση, έρευνα και ε, περισσότερη επένδυση σε αυτά, να παραμεριστούν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και βεβαίως οι προπολογισμοί να είναι προσανατολισμένοι προς το μέλλον. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί η Τραπεζική Ένωση, να έχει ουσία το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αυτά τα οποία ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης να εφαρμοστούν όσον αφορά τη δημοκρατική νομοποίηση, τον έλεγχο και τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Πρέπει τα μέτρα να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο και να σταματήσει επιτέλους αυτό το δράμα που βλέπουμε να Ευχαριστώ κύριε Κάρας. Ε, Η κυρία Μπερέζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη βυθίζεται όλο και πιο πολύ προς τον αποπληθωρισμό στην έλλειψη αναπτυξής και δεν κάνετε τίποτα. Η Κεντρική Τράπεζα αντέδρασε. Ο Μάριο Ντράγκη που θα θέλαμε να είναι μεταξύ μας σήμερα κατά κάποιον τρόπο έκανε μια αξιολόγηση της δράσης της Κομισιόν και την επέκρινε για τον τρόπο που αντιδράει. Τι λέτε λοιπόν εσείς γι' αυτό. Ακόμα περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι μια πραγματική διαρθρωτική μεταρρύθμιση πρέπει να επιτρέπει και στο ανθρώπινο κεφάλαιο να ζει. Εσείς κύριε Κατάινεν πώς προετοιμάζετε λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής με τα νέα στοιχεία και με τους αριθμούς του ΩΣΑ πότε θα αντιδράσετε για να κινητοποιηθεί η δυνατότητα που υπάρχει της εσωτερικής ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε θα αντιδράσετε για να εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα των 300 δισεκατομμυρίων που μας υπόσχονται και που θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση στην Ευρωζώνη για να δημιουργήσει μεγαλύτερη απασχόληση και περισσότερη ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερέσο. Ο κύριος Γκουερέρο. Λίγο πριν την Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά είχε δείξει ότι είναι πολύ ικανοποιημένη όπως το κάνει συχνά από τον εαυτό της. Είχε πει ότι τότε είχαμε βγει από την κρίση. Είχε τελειώσει η κρίση. Τώρα όμως από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μια τρίτη περίοδο ύφεσης. Η ανάπτυξη δεν είναι αυτή που περιμέναμε, για τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες επίσης της ζώνης ευρώ ισχύει το ίδιο. Γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς έχουμε μετατρέψει την ευρωπαϊκή οικονομία σε έναν χρόνιο θα έλεγα ανάπηρο μια κατάσταση με ε, επιβράδυνση των επενδύσεων, με μείωση των αμοιβών με υπερβολική λιτότητα καταστροφική. Λοιπόν, απαιτείται αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι το οποίο να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από την παιδεία, μέσα από τις επενδύσεις, μέσα από την ανάκτηση ε, των αμοιβών και των μισθών. Δεν ανήκουμε στους φίλους ε, της, ε, των ελλημάτων, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση σε σχέση με τη μείωση της ζήτησης είναι καρπός της πολιτικής που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Χωρίς ε, τις ερωτήσεις, χωρίς συγγνώμη επενδύσεις δεν θα υπάρξει ανάπτυξη, θα συνεχιστεί η φτώχεια και θα δημιουργούμε μια μάζα ε, εργαζομένων οι οποίοι θα ζουν στην ουσία μέσα σε συνθήκες ένδυας. Ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. Περνάμε λοιπόν τώρα στην διαδικασία του Catch the Eye. Έχουμε ένα πρόβλημα όμως. Έχουν ζητήσει 14 άτομα τον λόγο, 14 συνάδελφοι, φυσικά και δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε στους 14 το λόγο. Θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε λοιπόν στους χρόνους και γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας να μένει ε, στον χρόνο τον οποίο θα έχει στην διάθεσή του. Θα δώσουμε πάντως σε εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων τον λόγο έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιος αποκλεισμός. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι δεν είναι άσχημα τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ντράγκη, αλλά αυτό δεν αρκεί, λέει ο κύριος Σουσάλμπα Μπιντεγκάιν. Δεν θα λύσουν τα προβλήματα. Ε, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάρουμε μέτρα για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσουμε επιτέλους οικονομική ανάπτυξη. Η Ισπανία είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας μεταρρυθμιστικής είναι μια χώρα η οποία έχει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Αυτό όμως δεν αρκεί. Βρισκόμαστε παρά μόνο στην αρχή. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα παράδειγμα. Κύριε Επίτροπε λοιπόν, όχι μόνο θέλουμε μεταρρυθμίσεις, αλλά θέλουμε επίσης την εφαρμογή του προγράμματος του Juncker. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακούμε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν βλέπουμε συγκεκριμένα ίχνη του. Θέλουμε την απλή εφαρμογή του προγράμματος του Ιούνκερ. Ευχαριστώ κύριε Σάλμπα. Ο κύριος Μπαγιέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι η λεγόμενη έξοδος από την κρίση καταλήγει σε μια οικονομική ανάπτυξη 0%. Νομίζω ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη και μια αναθέρμανση θα ε. και δημόσιες επενδύσεις μαζικές και ελεγχόμενες. Ο κύριος Γιούνκερ μας υποσχέθηκε 300 δισεκατομμύρια για πρόγραμμα επενδύσεων και ο κύριος Δράγκη μας μίλησε για καλύτερη χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος να ανταποκριθούμε στην ε, διάσκεψη είναι να λύσουμε αυτά τα δύο προβλήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη. Γιατί αν δούμε τα πράγματα από κοντά βλέπουμε ότι όλα τα πρότυπα του Eurostat καταλήγουν στο ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνονται ιδίω στην πραγματικότητα των τοπικών κοινοτήτων και πρόκειται για λάθη. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, απογοητεύτηκα από αυτά τα οποία άκουσα. Εδώ και πέντε χρόνια τα ακούω αυτά και σε πέντε χρόνια πάλι τα ίδια θα μας λέτε. Καμία πρόοδος. Δεν ξέρω, είναι τυφλή η Κομισιόν. Στην πραγματικότητα ο κύριος Μαρόζο μας είπε πως η κατάσταση είναι καλύτερη από το 2010. Το αντίθετο ισχύει. Αυξάνεται τραγικά η ανεργία. Τα χρέη επίσης, η ανταγωνιστικότητα καθόλου από την άλλη πλευρά. Η δε ε, μας ε, ανέλησε την πολιτική της ενώπιων ε, νομπελιστών οι οποίοι πραγματικά την ε, εξευτέλισαν, της είπαν πως ε, η πολιτική σας οδηγεί στο τελείως αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο θέλετε. Δεν μιλήσατε καθόλου για ένα πρόγραμμα επενδύσεων. Επιτέλους οι χώρες πρέπει να μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο είναι προς το συμφέρον τους. Όσο έχουμε ευρώ τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα μέτρα τα οποία ζητάμε κάθε φορά να παίρνουν σε αυτές τις συναντήσεις πρέπει να εξυπηρετούν κάποιες κοινέ ιδέες, να προωθούν τα κοινά δίκτυα και ε, δεν θα πρέπει να περάσουμε σε, και να πέσουμε σε μια πολιτική διακυβέρνηση οικονομική της Ευρώπης καλύτερη με ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και δεν αρκεί εμείς να προσπαθούμε να παραμένουμε πάντα στις επιτυχίες τις οποίες σημειώσαμε τα τελευταία χρόνια. Απαιτούνται νέες επενδύσεις σε υποδομές, στις μεταφορές, Νομίζω επίσης ότι χρειάζονται και αρκετά μέτρα ε, σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό για τον κοινωνικό τομέα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν επιδεικνύουμε την απαραίτητη ε, ικανότητα να διαχειριστούμε τα πράγματα. Αν συνεχίσουμε έτσι τότε θα χάσουμε ακριβώς αυτό που είπατε κι εσείς, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Φερέιρα, η κυρία Φερέιρα. Όχι, ο κύριος Φερέιρα διορθώνει ο πρόεδρος. Αλλά δεν είναι στην αίθουσα ο κύριος Φεράρα, ο κύριος Ουρτασούν. Κύριε Κατάιναν, ε, υπάρχουν ε, από το προηγούμενο καλοκαίρι καταστροφικές, ε, θα έλεγα καταστροφικά στοιχεία λόγω ακριβώς της συνδυασμού αυτών των μεταρρυθμίσεων και της λιτότητας. Εσείς αυτό το οποίο μας ζητάτε κύριε Κατάινεν είναι να επιταχύνουμε την πορεία μας προς τον κρυμνό. Δεν είναι λογική αυτή, ιδιαίτερα για χώρες της περιφέρειας όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα κτλ. και θέλετε και η Ιταλία να κάνει το ίδιο. Να μειώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων μειώνοντας τις δημόσιες δαπάνες και να αφήσουμε ταυτόχρονα την οικονομία των καζίνο και να αφήσουμε τα χρήματα στα χέρια των αυτών οι οποίοι παίζουν με τα οικονομικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, πρέπει να ζητήσετε συγνώμη για τα προβλήματα που έχετε δημιουργήσει και τη δυστυχία που έχετε δημιουργήσει. Γιατί αλλιώς δεν μας είπατε τίποτα και δεν μας δώσατε καμία πληροφορία. Αναγνωρίστε τα λάθη σας και αλλάξτε την πορεία προς την αυτοκτονία. Ο κύριος Φερέιρα έχει επανέλθει και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εκλογές τελείωσαν και κάποιοι λένε πως τελείωσε και η κρίση στην Ευρωζώνη. Ε, και όμως τα πράγματα χειροτερεύουν στην πραγματικότητα. Και έχουμε δύο επιλογές, είτε τα ίδια και τα ίδια και βλέπετε πως ε, η Κομισιόν και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αυτό θέλουν ή αλλαγή. Αλλαγή μέσω μιας πραγματικής συζήτησης για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλαγή του καταστατικού της. Να μην ε, έχει πλέον ανεξαρτησία, να έχουν ξανά αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη για την νομισματική τους πολιτική. Αλλιώς θα έχουμε στασιμότητα. Πρέπει να ε, ε, έχουμε μια πραγματική λύση. Δεν γίνονται αυτά με ενιαίο νόμισμα. Έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά βλέπουμε που οδήγησε αυτό. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν ξανά τις εξουσίες τους. Σας ευχαριστώ. Έθριτς. Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για την οικονομική ανάπτυξη. Είτε πιστεύει κανείς πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη είναι κάτι καλό, είτε θεωρεί κανείς όπως εγώ ότι είναι κάτι το αποτρόπαιο. Αλλά όλοι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να γίνει με το να απελευθερωθούν οι λαοί της Ευρώπης από τις αλυσίδες που τους κρατάνε και αυτές είναι το υπερβολικό κράτος, η υπερβολική φορολογία που τους περιορίζουν. Ελευθερώστε την επιχειρηματικότητα των Ευρωπαίων για να δουλέψουν μέσω του, της δικής τους δημιουργικότητας να μπορέσουν ξανά να δημιουργήσουν. Απευθύνω έκκληση ειδικά στην Κομισιόν σκεφτείτε αυτές τις ιδέες. Όλοι θέλουμε να είμαστε καλύτερα, με περισσότερη ευημερία και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δημιουργικότητά μας για να το επιτύχουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Έθριτς για την Κομισιόν ο κύριος Κατάινεν. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, και εγώ θα ήθελα περισσότερη συζήτηση μαζί σας, αλλά πρέπει να φύγω σε αποστολή σε λίγες ώρες. Ο κύριος Μπάλτ υπενθύμησε ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται με στόχο να αυξήσουν την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη. Πολύ σωστό. Δεν έχουμε μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειάζονται διάφορες μεταρρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα. Δεν χρειάζονται οι ίδιες σε κάθε χώρα. Εξαρτώνται πολλές φορές από την τοπική κατάσταση. Εύκολο είναι να συμφωνήσω με την κυρία Ροντρίγκε που είπε ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και επίσης υπενθυμίσατε την ανάγκη οι μεταρρυθμίσεις να ενδυναμώνουν την καινοτομία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να οργανώσει κανείς να διαχειριστεί την καινοτομία στις χώρες μέλη και εμείς θέλουμε να εμπνευστούμε από τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στις διάφορες χώρες γιατί αυτό θα μπορούσε να ανανεώσει την Ευρώπη. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις μας προχωράνε. Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία στην Ευρώπη αλλά και μερικές αδυναμίες και ελλείψεις και εγώ προσωπικά πιστεύω στην έρευνα και την καινοτομία. Καινοτομία σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλη, θα δίνεται μεγάλη σημασία στην έρευνα και στην επιχειρηματικότητα. Τίθεται όμως το πρόβλημα του πώς να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι δημόσιοι πόροι που διαθέτουμε. Um, um, Η ΕΤΕ θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτό. Και είπατε και πολλοί από εσά ότι είναι σημαντικό οι επενδύσεις να μην γίνονται τυφλά. Οι επενδύσεις όμως σημαίνουν ζήτηση, σημαίνουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη και γι' αυτό πρέπει να συνδυάσουμε τις μεταρρυθμίσεις με περισσότερη ζήτηση και δημοσιονομική πειθαρχία και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Η Κομισιόν, η νέα Κομισιόν ή μάλλον οι νέοι επίτροποι, υποψήφοι επίτροποι, θα προσπαθήσουν να τα καθορίσουν όλα αυτά στις προγραμματικές τους δηλώσεις. Σε άλλη φορά θα τα πούμε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Επίτροπε και τώρα για το Συμβούλιο ο κύριος Δελαβέντοβα για να συνοψίσει. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα την οποία δώσατε στην Προεδρία να ακούσει μια ευρυτάτη παρουσίαση των απόψεών σας. Οι παρεμβάσεις σας ξεπέρασαν πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα της συνάντησης κορυφής της ζώνης ευρώ που θα γίνει τον επόμενο μήνα αλλά όπως σας είπα δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτό σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα εξ αρχής. Να επαναλάβω όμως ότι θα είμαι σε θέση να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όταν συγκληθεί επισήμως η συνάντηση αυτή στην επόμενη ολομέλειά σας. Ε, σε σχέση με τις ε, προθεσμίες, τις χρονικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις και τα λοιπά, στα οποία αναφερθήκατε να επαναλάβω ότι η Ιταλική Προεδρία, επαναλαμβάνω, έχει σαν βασική προτεραιότητα και σαν κατεπήγον θέμα τον χρόνο με τον οποίο θα τεθούν σε εφαρμογή οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν. Και συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι σημείωσα προσεκτικά όλα όσα μας είπατε και τις προτάσεις σας και θα προσπαθήσουμε οι προτάσεις αυτές, οι συστάσεις αυτές να μεταφερθούν σε όσους εμπλέκονται στην προετοιμασία της επόμενης συνάντησης κορυφής της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαριανόπουλο για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, στην διάρκεια της διαδικασίας δόθηκε ο λόγος σε κάποιον συνάδελφο ως ε, εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων ε, βουλευτών. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι πολύ καθαρός. Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν αποτελούν, δεν αποτελούν πολιτική ομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν ενιαία πολιτική έκφραση, άρα κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Ο καθένας τοποθετείται ανάλογα και εκ μέρου του εθνικού κόμματο με το οποίο έχει εκλεγεί σε αυτή τη Βουλή. Άρα το σωστό όταν δίνεται ο λόγος σε μία εγγεγραμμένο βουλευτή θα ήταν ότι δίνεται ο λόγος στο μία εγγεγραμμένο βουλευτή τάδε ονόματο. Αυτά σας ευχαριστώ. Thank you for that point of order and we will take note of your comments. Um, θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας. Τώρα περνάμε ε, στην ε, δήλωση, στη συζήτηση για την εκκίνηση της πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Νεότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα ε, θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σεβαστείτε όσοι σηκώνετε την μπλε κάρτα τα 30 δευτερόλεπτα για να υπάρξουν 20 με 30 δευτερόλεπτα για απάντηση.